Witam Państwa. Ευχαριστώ. Έχω τώρα την τιμή να ε, συνεχίσω να προεδρεύω κατά τη διάρκεια των ε, επεξηγήσεων ψήφου. Περιμέναμε λίγο για να παραμείνουν όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν το λόγο και να ακούσουν και οι υπόλοιποι να αποχωρήσουν. Ε, θυμίζω σε εκείνους που έχουν παραμείνει στην αίθουσα και θέλουν να μιλήσουν ότι ε, εδώ έχουμε επεξηγήσει ψήφου και παρακαλούνται οι ιδιωτικές συνομιλίε εκτός τη αιθούση να συνεχιστούν. Λοιπόν, έχουμε τώρα την έκθεση του κυρίου Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες και του κυρίου Μπούλμαν με θέμα την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Πέντε συνάδελφοι παρακάλεσαν να τους δοθεί ο λόγος για επεξήγηση ψήφου. Πρώτος, ο κύριος Μόμτσιλ Νέκοφ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων ήδη ε, λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. Όμως βλέπουμε να υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Τον Ιούλιο του 2016